So good afternoon, ladies and gentlemen. May I just draw your attention just for a couple of minutes of housekeeping points. Παρακαλώ να ξεκινήσω με κάποια διαδικαστικά όσο περιμένουμε να έρθει ο Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Παπαδημούλη, για να κηρύξει επισήμω την έναρξη των εργασιών τη ημερίδα αυτή. Θέλω να σα καλωσορίσω σε αυτό το σεμινάριο τύπου που οργανώνουμε επ' ευκαιρία τη Διεθνού ημέρας τη Γυναίκα. Εγώ θα είμαι ο σύνδεσμος ε, και ό,τι θέλετε και στο κοκτέιλ. Ρίξτε τα όλα πάνω μου. Ε, αν έχετε κάποια παράπονα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα το αντιμετωπίσω. Τρεις μήνες μας μένουν από τις ευρωεκλογέ από την 5η 23 έως ε, την ε, Κυριακή 26 Μαΐου και η ισχύ των γυναικών είναι το θέμα μας. Κάποια πρακτικά να σας πω. Βλέπετε τις καμπίνες διερμηνίας. Συνάδελφοί μας διερμηνείς θα σας παράσχουν διερμηνίες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ελληνικά. Από και προς. Αύριο θα έχουμε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πολωνικά και πορτογαλικά. Έχετε λάβει το φάκελο τύπου. Φαντάζομαι αύριο θα σας ε, διανύμω και μια εργαλειοθήκη. Ε, βλέπετε τον κωδικό για το Wi-Fi στην έσοδο. Και επίσης ε, ελεύθερα φωτογραφίστε ό,τι θέλετε και μπορείτε να αποστάρετε στα κοινωνικά δίκτυα τις φωτογραφίες αυτές. Επίσης υπάρχει ζωντανή μετάδοση του σεμιναρίου στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου. Μπορείτε να στείλετε την ηχογράφηση και τη μαγνητοσκόπηση στους κοινωνικά μέσα επίσης. Θα στείλω αύριο ένα email και θα σας ε, δώσω όλο το ακουστικό περιεχόμενο, της θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όταν ε, κάνετε τα ρεπορτάζ σας για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας. Κάτι σημαντικό, παρακαλώ, να υπογράψετε ε, την, το παρουσιολόγιο σήμερα και αύριο. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να σας επιστραφούν τα έξοδά σας. Παρακαλώ λοιπόν να γράψετε, τα, να υπογράψετε. Will be back to... Οι συνάδελφοί μου ε, θα είναι εδώ από το Reimbursement Desk και αν λείπει κάτι από τις 8.30 μέχρι τις 9.30 αύριο το πρωί μπορείτε να τους ε, συναντήσετε και πάλι και να δώσετε τα έγγραφα, τα αποδεικτικά. Αν όχι, στείλτε τα παραστατικά ταχυδρομικά. Μην ε, δηλαδή σας πιάσει και άγχος και με αυτό για τις συνεντεύξεις. Κάποιοι έχετε ζητήσει συνεντεύξεις με μέλη του πάνελ. Αυτές οι συνεντεύξεις θα γίνονται στην είσοδο. Υπάρχει ένας χώρος εκεί και με κάποιους καναπέδες. Όποιοι έχετε ζητήσει συνεντεύξεις, αν υπάρχει δυνατότητα θα σας ε, καλύψουμε όλους. Αλλά θα δώσουμε προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν ήδη ζητήσει να κάνουν κάποια συνέντευξη. Σήμερα το μεσημέρι ε, υπάρχει δυνατότητα να έρθετε σε επαφή με τους συναδέλφους σας στη διάρκεια του κοκτέιλ που θα ακολουθήσει. Οι συνάδελφοί μου και εγώ θα σας δείξουμε που είναι στο κτίριο Γιώζεφ Αντάλ στον τρίτο όροφο. Το έχετε το όνομα Μπρασέρι λέγεται, αλλά θα σας ε, οδηγήσουμε εμείς μετά τη λήξη της απόψινής συνάντησης στο χώρο αυτό. Και κάτι τελευταίο, έχετε για σήμερα και για την πέμπτη διαπίστευση. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε κάποια συνεδρίαση ε, συγκεκριμένα την Επιτροπή Γυναικών, οπότε κρατήστε ε, τη διαπίστευση για να μπορέσετε να μπείτε χωρίς τη δική μας βοήθεια αύριο. Σε οποιαδήποτε είσοδο, αν πάτε, θα μπορέσετε να μπείτε. Εδώ θα ε, να συνεδριάσουμε αύριο και για την Επιτροπή Γυναικών την Πέμπτη. Μπορείτε να δείτε σε ποια αίθουσα συνεδριάζει η Επιτροπή Γυναικών, μπορείτε να πάτε και εκεί. Αυτό το σεμινάριο στόχο έχει να συνεισφέρει στη συζήτηση κυρίω για την ισότητα των φύλων, τι γυναίκε σε θέση ισχύω, εν των ευρωεκλογών του Μαΐου. Περιμένουμε και ελπίζουμε να βρείτε επικοδομητικό και χρήσιμο για τα ρεπορτά σα ε, το σεμινάριο αυτό. Και τώρα έχω τη χαρά να δώσω το λόγο σε έναν από τις συναδέλφους σας, ε, την Τερέσα Κιούχλερ, ε, που είναι ανταποκρίτρια ε, στη σουηδική εφημερίδα Dag Bladet. Θα είναι η συντονίστρια σήμερα και αύριο. Έχει την άντρες εδώ στις Βρυξέλλες. Τερέσα, ορίστε, έχεις το λόγο. Καλώς ήρθατε. Δεν βλέπω καθόλου Σουηδούς στον κατάλογο. Υπάρχει κάποιος Σουηδός. Όχι, είμαι η μόνη Σουηδέζα στην αίθουσα. Καλώ ήρθατε. Ήμουνα και πέρυσι ε, ε, και συμμετείχα σε ένα από τα πάνελ. Ε, πέρυσι ε, ήταν η συνεδρίαση αυτή μετά από την σύμπηξη του κινήματος MeToo. Ε, Υπήρχε και μεγάλη απογοήτευση. Πολλές γυναίκες μιλούσαν για τις εμπειρίες τους με την ε, παρενόχληση, αλλά κάναμε και brainstorming, συζητήσαμε για το πώς αντιμετωπίσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο εδώ το, το θέμα της παρενόχλησης. Ε, όχι εγώ προσωπικά, εντάξει, αλλά και οι δημοσιογράφοι. Ε, και φέτος θα υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον ε, εν ώψη των ε, επικείμενων ευρωεκλογών, λιγότερο από 100 μέρες μας μένουν. Ε, τα πάθια να βράζουν εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία φέτος για να θέσουμε κάποια θέματα για την ισότητα των φύλων. Ε, ξέρετε ότι οι πολιτικοί θέλουν να προσελκύσουν ψηφοφόρους. Δεν νομίζω ότι η συζήτηση για τα γυναικεία θέματα θα είναι λιγότερο ε, έντονη. Ελπίζω λιγότερο φλιβερή πάντως. Θα έχουμε δύο μέρες μπροστά μας με πολιτικούς, ε, είμαι έτοιμη για μάχη μαζί τους. Θα κάνουμε θα, κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις, τι κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στον τομέα της ισότητα των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, τι κάνουν για την παρενόχληση. Ε, ο βασικός μας ομιλητής διαρωτώ αν έχει φτάσει ήδη, θα κάνει τη βασική παρουσίαση, θα έρθει όπου να είναι. Να σας πω δύο λόγια εγώ τότε από πλευράς μου. Αυτή η διάσκεψη δεν είναι αυτή η κυρία που μπήκε. Φέτος αυτή η διάσκεψη λοιπόν γίνεται δύο μέρες πριν από την ε, μέρα της γυναίκας. Η 8η Μαρτίου είναι η μέρα που δεν είναι αργία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πέρυσι ήταν η Ευρωπαϊκή ημέρα στις 8 Ιουνίου, αν δεν απατώμε, για την Ευρώπη. Σωστό δεν είναι αυτό που λέω. Ναι, η 8 Ιουνίου. Και συζητούσαμε το γιατί προωθούμε την ιδέα της αργίας για την 8η Μαρτίου. Ξέρετε τι γιορτάζουμε σε 8 Μαΐου, διορθώνει Μιλίτη, όχι 8 Ιουνίου. Ξέρετε τι γιορτάζουμε. Ένα άτομο γνέφει. Εσείς που γνέφετε, ξέρετε τι γιορτάζουμε την 8η Μαΐου. Είναι μια συγκεκριμένη δήλωση αυτή που γιορτάζουμε, τη δήλωση Σούμαν. Κανένα δεν το ήξερε, ούτε εγώ το ήξερα. γιατί συζητούσαμε γιατί έχουμε αργία 8 Μαΐου. Ε, εμείς προωθούμε λοιπόν και την 8η Μαρτίου ως ε, ημέρα αργίας. Θα μας πει δύο λόγια όταν έρθει για το τι κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τα θέματα γυναικεία. Okay. Okay.